Meine Κυρίες αλλά και κύριοι, καλώς ήρθατε στην κοινή συνεδρίαση της ΑΦΕΤ και της ΕΝΒΗ, μαζί με τον κύριο Λαβία, ο οποίος θα συμπροεδρεύσει. Δεν βλέπω ακόμα την κυρία Πιετικάινεν, και καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορέσει να παρασταθεί στην συνεδρίασή μας, αλλά ο κύριος Πέτερ Λίζε θα την αντικαταστήσει. Βέβαια, δεν θα μπορέσει να παραμείνει πάρα πολύ ώρα στη συνεδρίασή μας. Αν συμφωνείτε λοιπόν κύριε Λαβία, μπορούμε να δώσουμε κατευθείαν τον λόγο στον κύριο Πέτερ Λίζε. Και γι' αυτό και εγώ ίδιος δεν θα κάνω τώρα μακρά παρουσίαση και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον Πέτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι χρειάζεται να αντικαταστήσω την κυρία Πίντι η οποία ζητά συγγνώμη για την απουσία της. Είχε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα και επομένως αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει στην ε, στην, ε, στην εκλογική της περιφέρεια. Εγώ φυσικά είμαι εδώ για να παρουσιάσω την άποψή της και θα καταγράψω όλα αυτά τα οποία θα πούν οι συνάδελφοι και φυσικά θα τις θα διαβιβάσω στην κυρία Πίτη Κάινεν. Κάτι το οποίο μπορώ να πω ήδη προσωπικά είναι ότι εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν είμαστε ιδιαίτερα πολυπληθής, αλλά αυτό μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κοινέ συνεδριάσεις και στα πλαίσια της συνεδρίασης, της συνδιάσκεψης που γίνεται για την κλιματική πολιτική, να μπορέσουμε να συνδυάσουμε <clears throat> τις ενέργειές μας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια είναι στα αγγλικά τώρα τα, τα, οι σημειώσει της κυρίας Πιετικά και θα τα διαβάσω στα στα αγγλικά, στα φιλανδικά, στα φιλανδικά λέει ο πρόεδρος. Α, δεν είναι πολύ καλά τα φιλανδικά μου. Θα προσπαθήσω στα αγγλικά. Καταρχήν η κυρία είναι, θέλει να συγχαρεί την Κομισιόν για την εξισορροπημένη ε, κατάληξη στην οποία φτάνει η ανακοίνωση από την Κομισιόν και την ύπαρξη εκπρόσωπο σε σχέση με την ακτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι είναι μια καλή βάση για την ανάπτυξη μιας αρχικής διάστασης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης θέλει να ευχαριστήσει την Επιτροπή ΑΦΕΤ και τον συνεισηγητή της τον κύριο Πατ, αν το προφέρω σωστά, και χαίρεται για την πολύ καλή συνεργασία που είχε από τον συνεισηγητή τη για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για την ακτική. επομένω θα πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία της εκεί τα ανθρώπινα θέματα, τα θέματα περιβάλλοντος, τα θέματα ασφάλειας ακτικής, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την σταθερότητα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να θέσουμε στο προσκήνιο τις προκλήσεις για το περιβάλλον για το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κλιματική αλλαγή γίνεται πιο γρήγορα στην Αττική από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου μας. Αυξάνει η θερμοκρασία, ε, λιώνει ο ακτικός πάγος και αυτό θέτει τον κίνδυνο αύξησης του επίπεδου της θάλασσας. Αλλάζει και η σύνθεση των υδάτων και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε απρόπτα κλιματικά σχήματα και μορφές καιρού. Όλα αυτά λοιπόν δεν επηρεάσουν μόνο τις χώρες της Ακτικής, αλλά όλες τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε εύκρατα κλίματα. Η ρήπανση στην Ακτική προέρχονται κυρίως από την Ασία, την ε, Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Επομένως, τα μέτρα μείωση των εκπομπών από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξουν σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη κλιματική αλλαγή στην Αρκτική. Θα πρέπει οι βιώσιμοι στόχοι του για, το, για την ανάπτυξη να αντανακλώνται καλύτερα στην Αρκτική, όχι μόνο γιατί όλε οι χώρε μα έχουν δεσμευτεί να μπορέσουν να επιτύχουν αυτού του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά επίση είναι ιδιαίτερα εύθραστή η φύση στην Ακτική και χρειάζεται ένα ενισχυμένο επίπεδο υποστήριξης και προστασίας. Η βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν είναι η μόνη μορφή ανάπτυξη η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Ακτική περιοχή και επομένω η πολιτική μας για την Ακτική θα πρέπει να αντανακλά καλύτερα τις απαιτήσει των βιώσιμων στόχων ανάπτυξη μέσα στην περιοχή αυτή με ιδιαίτερη <clears throat> εστίαση στη διατήρηση των οικοσυστημάτων οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη μα δίνουν το σωστό πλαίσιο για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στην ικανότητα του οικοσυστήματο που υφίσταται πιέσει από αρνητικέ επιπτώσει ε, στο περιβάλλον που επιταχύνονται και από την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να προστατευτεί καλύτερα η φύση τη ακτική με το να έχουμε ειδικέ για την ακτική μελέτε αντικτύπου. Αυτό θα βοηθήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει με πιο υπεύθυνο τρόπο και να χρησιμοποιήσει καλύτερα τους πόρους που προερχόνται από την περιοχή της Ακτικής. Μια σωστή λοιπόν <clears throat> αντιμετώπιση θα πρέπει να περιλαμβάνει και καλύτερους μηχανισμούς διαβούλευσης και συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών. Προτείνει η κυρία Πιέτη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπενθυμίσει και πάλι την αίτησή του από το 2011 να απαγορευτεί η χρήση βαρέων ε, κλασμάτων πετρελαίου στην Αρκτική, κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί στην Αντακτική. Γιατί υπάρχουν κίνδυνοι από τρει μορφέ τριών ειδών. Οι απορρίψει πετρελαίου, οι διαρροέ και ο κίνδυνο για την περιοχή αυτή, μετά ο μαύρο άνθρακο, ο άνθρακο δηλαδή σε μικροσωματίδια που έχει αρνητικά αποτελέσματα και επιταχύνει την τήξη των πάγων και του χιονιού. Η κυρία Πετικάνη χαιρετίζει την πρόταση της Κομισιόν όταν υπογραμμίζει την ανάγκη να πάρει πρωτοποριακό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της έρευνας και πιστεύει ότι μπορούμε να έχουμε ένα, μια αποστέμενη αξία στον ερευνητικό τομέα για την Αρκτική και επομένως θα πρέπει να, συνε, να διατηρηθούν τα κονδύλια έρευνας και για το επόμενο διάστημα προγραμματισμού. Με καλύτερη συνέχεια και καλύτερο συντονισμό της έρευνας <clears throat> μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και η έκθεσή της Τονίζει και πάλι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει ένα κέντρο πληροφορία για την Ακτική για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τη περιοχή. Αυτά θέλησε η κυρία Πιετικάινεν να σα μεταφέρω. Λυπάμαι και εγώ που δεν μπόρεσε να είναι παρούσα η κυρία Πιετικάινεν και εγώ θα πρέπει να φύγω σύντομα για μια άλλη συνεδρίαση. Αλλά είναι εδώ και ο βοηθό τη κυρία Πιετικάινεν ο οποίο θα καταγράψει τι ε, σα και θα μεταφέρει οποιαδήποτε ερωτήματα στην ε, εισηγήτρια και φυσικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε και την άποψη του συνεισηγητή από την Επιτροπή ΑΦΕΤ και όπως και όλων των άλλων συναδέλφων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρόκ και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ για την ε, κοινή αυτή συνεδρίαση και την επικοδομητική συνεργασία που έχουμε ανάμεσα στις δύο επιτροπές μας. Είναι πολύ σημαντικό μέσω της έκθεσης αυτής να καταφέρουμε να προστατεύσουμε την ικανότητα του οικοσυστήματος της Αρκτικής. Προσβλέπω λοιπόν στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε σήμερα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε τώρα να ακούσουμε τον εισηγητή από πλευράς ΑΦΕΤ, τον κύριο Ούρμα Σπάιτ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε όλοι, η γεωπολιτική σημασία της περιοχής Αρκτικής αυξάνεται όλο και περισσότερο. Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, καθώς επίσης και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για την πρόσβαση στους πόρους της Αρκτικής και στις οικονομικές δραστηριότητες εκεί, φέρουν τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις όμως για την όλη περιοχή. Περιλαμβάνονται λοιπόν κάποιες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, καθώς μεταμορφώνται όλο και περισσότερο η οικονομική δραστηριότητα στην Αρκτική. Η Αρκτική όλο και περισσότερο ήταν μια περιοχή επικοδομητικής συνεργασίας και έχει παραμείνει μια περιοχή όπου υπάρχουν χαμηλές τελικά εντάσεις και περισσότερο έντονη συνεργασία. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να διατηρηθεί. Είναι σημαντικό να παραμείνει η αρκτική περιοχή χαμηλών εντάσεων. Υπάρχει μάλιστα εκτεταμένο διεθνές νομικό πλαίσιο που ισχύει για την Αρκτική και στα πλαίσια αυτού του πλαισίου διευθετούνται όλα τα ζητήματα κυριαρχία στην Αρκτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει στην Αρκτική μακροχρόνια δράση, η οποία βασίζεται στην ιστορία, στη γεωγραφία, στην οικονομία και στην έρευνα. Τρία κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δανία, η Φιλανδία και η Σουηδία, είναι πλήρη μέλη του Οκτωμελού Αρκτικού Συμβουλίου και άλλα επτά κράτη-μέλη είναι παρατηρητέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει όμω ακόμη να τη χορηγηθεί καθεστώ παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο. Και καθώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριο χρηματοδότη στην Αρκτική, θα ήταν απόλυτα εύλογο να αναβαθμιστεί το καθεστώ τη στο Αρκτικό Συμβούλιο και να γίνει παρατηρητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρτήσει και ενισχύσει σταδιακά την πολιτική τη για την Αρκτική. Έχουμε την κοινή ανακοίνωση τη Επιτροπής καθώς επίσης και την παγκόσμια στρατηγική που αναφέρεται στην πτυχή ασφάλειας για την Αρκτική. Οι γεωπολιτικέ εξελίξει στην περιοχή τη Αρκτική επηρεάζουν επίση την κατάσταση ασφάλεια στη Βόρεια Ευρώπη αλλά και παντού στον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώ τον, κόσμο, τον, τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε οποιαδήποτε αστρατικοποίηση στην Αρκτική. Γι' αυτό ακριβώ και στην έκθεση λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εσωτερικέ και εξωτερικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στρατηγική για την Αρκτική και να αρχίσει να δεσμεύεται όλο και περισσότερο Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σημαντική αυτή περιφέρεια, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι πτυχέ. Η ανάγκη αυτή προκύπτει μεταξύ άλλων και από το γεγονό ότι όλα τα αρκτικά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα άλλα κράτη έχουν τι δικέ του εθνικέ στρατηγικέ για την Αρκτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ικανότητα να συμβάλλει με πολλαπλού τρόπου στην αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων, για την ασφάλεια και την αποτροπή των συγκρούσεων και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη τη στη δημιουργία μηχανισμών για την ασφάλεια των πολιτών καθώ και στη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και των υποδομών έρευνα και διάσωση. Η έκθεση ζητεί μια βιώσιμη πολιτική για την Αρκτική και φυστά την προσοχή στο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί απαραίτητο το σεβασμό του διεθνού δικαίου στην Αρκτική και τάσεται υπέρ ενό ισχυρού ρόλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόθεση αποτελεσματικών πολυμερών ρυθμίσεων και μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνε. Θα ήθελα προφανώ να ευχαριστήσω και την ε, συνεισηγήτρια από την ΕΝΒΗ, την κυρία Πιέτη Κάινεν, θα συνεχιστεί προφανώς η εργασία μας και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα θετικό συμπέρασμα και ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε σε μια επόμενη ολομέλεια την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. No. Τώρα, ο κύριος Ντόνζον. Merci, Monsieur le Président. <clears throat> C'est mon collègue. Σας ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τον κύριο Μίκαλ Γκάλερ οποίο ήταν ο σκιώδη συζητητή για το θέμα αυτό, αλλά κολλείεται δυστυχώ και ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Έπρεπε να είναι παρόν σε μια συνδιάσκεψη για την πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Επομένω, θα μεταφέρω στα αγγλικά τι σημειώσει που μου άφησε για την έκθεση αυτή. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άμεσε απειλέ σε ό,τι αφορά την σταθερότητα τη Αρκτική. Υπάρχουν διάφορες περιοχές που αντίθετα μάλλον από άλλες περιοχές στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκεί είναι ένας χώρος ειρήνης και διεθνούς συνεργασίας και συμμετέχουν και μη κρατικοί φορείς. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ακτική εστιάζεται ιδιαίτερα στα θέματα του περιβάλλοντος και την επιστημονική έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει την οικονομική, οικονομικές δυνατότητες αλλά και τις πολιτικές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν από το να υπάρξει ελεύθερη πάγου διέλευσης στα ύδατα της Ακτικής. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Κομισιόν και της ΥΠΑ της για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και της πολιτικής για την ακτική των κρατών μελών μαζί με τις συνδεόμενες χώρες της Νορβηγίας και Ισλανδίας που θα οδηγήσουν και σε νέες πρωτοβουλίες. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν την ε, <clears throat> πρόταση να υπάρξει μια ομάδα εργασίας για την συνεργασία στον χώρο της Βόρειας Ευρώπης και τα θέματα της Ακτική. Χρειάζεται ένας πιο έντονο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ακτικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Από το 2012 και εντεύθεν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει επίμονα την ανάγκη να υπάρξει <clears throat> μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα των ε, φυσικών πόρων και της ασφάλειας για την περιοχή αυτή. Και εδώ πρέπει όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο Αρκτικό Συμβούλιο να δημιουργήσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για να αποφύγουν τις αντιπαραθέσεις για τους φυσικούς πόρους και να υπάρξουν και μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχομένων αντιπαραθέσεων. Επίσης, η παράγραφος 6 της ε, κοινή έκθεση πρέπει να υποστηριχθεί. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν πάντα ε, εκθέσεις για επιπτώσεις πάντα όταν γίνονται έργα στην περιοχή αυτή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση στην ε, περίπτωση της αυτή και επίσης 2 υπογραμμίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο και για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η θέληση σε πολιτικό επίπεδο να περιοριστεί η λειτουργία αυτή μόνο σε επιστημονικό επίπεδο. Έχουμε καταθέσει λοιπόν και μια σειρά τροπολογιών σε σχέση με όλα αυτά στην έκθεση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σαλτεμόζα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν δανέζικα και είχα προετοιμαστεί για τα δανέζικα. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, διευθυντές για την εξαιρετική τους έκθεση. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για την δουλειά μας και θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε πολλά ζητήματα. Εγώ είμαι σκιώδη ηγητρία των σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και ε, θα εστιάσω στα ζητήματα περιβάλλοντος. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε το ότι αυτό το οποίο γράφει η έκθεση, ότι πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην Αρκτική και συμφωνώ πλήρως ότι θα πρέπει ε, εφόσον είναι και μια περιοχή χαμηλών εντάσεων ε, μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα το περιβάλλον. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε και πρέπει να το γράψουμε στην έκθεση ότι η λήψη αποφάσεων για την Αρκτική θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με τους τοπικούς και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Θα ήθελα να πω ότι όταν μιλάμε για τις περιβαλλοντικές πτυχές ε, θα, θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσουμε τις ε, διατυπώσεις που υπάρχουν για να τονιστεί περισσότερο η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και βεβαίως να λάβουμε υπόψη τους ντόπιους και αυτόχθονες πληθυσμούς. Σας ευχαριστώ κύριε Φωτίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σκιωδησής ηγήτρια του ECR στην Άθλετ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Και ε, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκτιμώ ιδιαίτερα το κομμάτι της Envy ειδικά για επίσης και τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας που αναφέρει η Θα ήθελα να τονίσω εδώ την ε, πρόβλεψη υπάρχει την διάταξη για μια περιοχή χαμηλών και καθόλου ε, εντάσεων. Σωστά είπαν οι συνεισηγητές πως υπάρχουν τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές ε, στην θέση της Αρκτικής στις διεθνείς σχέσεις. Και δυστυχώς σε αντίθεση με τα όσα είχαμε προβλέψει και στα έγγραφά μας και στο διεθνές νομικό σύστημα, εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της περιοχής αυτής από την Ρωσική Ομοσπονδία. Απόδειξη αυτού είναι η λειτουργική αλλαγή εντός του ρωσικού στρατού που πλέον έχει μονάδες ε, για αυτήν την περιοχή ειδικά. Πρέπει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει ειρηνική συνεργασία σε όλους τους ε, τομείς συνεργασίας στην Αρκτική. Ε, είτε μιλάμε για το Συμβούλιο της Αρκτικής είτε για το Συμβούλιο της Θάλασσας Μπάρενς το Ευρωαρκτικό. Επίσης, ε, σημασία έχουν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών εκεί και άρα όλα τα διεθνή νομικά έγγραφα που αναφέρθηκαν στην αρχή της έκθεσης έχουν μεγάλη σημασία. Υπάρχει επίσης εδώ πέρα μια έκκληση για ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαίως αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης την παράδοση του καθεστώτος παρατηρητή ορισμένων χωρών όπως η Πολωνία που συνεισφέρουν πάρα πολύ. Και βεβαίως μιλάμε για την ε, ανάγκη συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του, των μελών του Συμβουλίου της Ακτικής, αλλά πρέπει επίσης να δούμε και τις εμπειρίες και τον ρόλο των κρατών μελών που είναι αυτή τη στιγμή παρατηρητές των προσπαθειών αυτών στην Αρκτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γετερμάκη. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω φινλανδικά, γιατί ο Έρμαρ Μπρόκ είπε ότι θα έπρεπε και ο σα να μιλούσε φιλανδικά. Ένας άλλος ομιλητής δηλαδή, που θα ακολουθήσω τη συμβουλή του. Ευχαριστώ λοιπόν Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συνσηγητές για την πολύ καλή αυτή έκθεση, το σχέδιο έκθεσης. Αναφερόμαστε πολύ στις κλιματικές αλλαγές και στην κατάσταση του περιβάλλοντος όσον αφορά την περιοχή της Αρκτικής. Υποστηρίζω εν γέννη το κείμενο. Θα ήθελα ωστόσο να υποβάλω και κάποιες τροπολογίες να κάνω μη άλλο κάποιες προτάσεις για να γίνουν κάποιες προσθήκες στο κείμενο. Πρώτον, είναι πολύ θετικό το ότι ε, αρχίζουμε και επενδύουμε όλο και περισσότερο στις ε, ευρωαρκτικές περιοχές. Οι δικές μας οι πολιτικές και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως γνωρίζετε στο παρελθόν επικεντρώνταν περισσότερο στην αρκτική περιοχή που βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικό και θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και περισσότερο επικεντρώνεται στο τμήμα εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην αρκτική περιοχή. Έχουμε αρκτικές ευρωπαϊκές περιοχές. Η συνεργασία λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αρκτικής είναι πολύ ψηλής ποιότητος είναι ιδιαίτερα επικοδομητική και όλοι οι παράγοντες στην περιοχή αυτή αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία αυτή είναι πολύ θετική. Είναι πολύ σημαντικό όμως και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίσει επισήμως ότι όντως δεν η συνεργασία στην περιοχή αυτή και έχοντας αυτό κατά νου θεωρώ ότι κάθε φορά που εξετάζουμε τη διατύπωση που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε μια τέτοια έκθεση θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι δεν θα συμβάλλουμε κι εμείς με τέτοιες εκθέσεις στην αύξηση της έντασης στην περιοχή, χρησιμοποιώντας λανθασμένες ή άκερες ή ατυχές εκφράσεις. Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των χωρών που βρίσκονται στον αρκτικό κύκλο είναι ότι, έχουν, ότι είναι περιοχές αεροκατοικημένες με ένα πολύ δύσκολο κλίμα ουσιαστικά, με πολλέ κλιματικέ αντικσότητε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν και επιθυμούν να ζουν σε αυτή την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και οι βόρειε αυτέ περιοχέ να συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο TNT, στο δίκτυο των αντιευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούμε περισσότερα έργα στην περιοχή αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε επίση στην περιβαλλοντική διάσταση των πολιτικών μα, αλλά να επιμείνουμε επίση και στη διάσταση εκείνη που έχει να κάνει με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Οι πολιτικές της βόρειας διάστασης επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε και στην περιοχή αυτή επιτυχείς πολιτικές και εταιρικές σχέσεις που είχαμε στον τομέα των μεταφορών ή στον ε, τομέα των logistics είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής αυτής να μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και να επιθυμούν όλο και περισσότεροι να ζουν σε αυτή την περιοχή. Είναι άλλωστε οι πολίτες αυτοί ισότιμοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Βαρέχο έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. φορές δεν έχουμε πραγματική συνείδηση του τι σημαίνει η περιοχή της ε, Οι βόρειες χώρες βέβαια της Ευρώπης ξέρουν ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της ε, επικράτειάς της και της κληρονομιάς τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη επίγνωση του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Αρκτική και πώς θα πρέπει να δράσουμε στον στο θέμα αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν πιο ψηλά από τον ακτικό κύκλο. Δεν είναι, δεν είναι πολλοί άνθρωποι, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι παρόλα αυτά χρειάζονται να έχουν καλύτερες υποδομές, ιδίως δυνατότητες επικοινωνία και συγκοινωνία. Ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο, στα βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλάμε όμω για την ακτική, εγώ σκέφτομαι πρώτα απ' όλα την ανάγκη να προστατεύσουμε την Αρκτική από εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της, να αποτρέψουμε την τήξη των πάγων της περιοχής αυτής και να έχουμε μια αντιμετώπιση διαφορετική για αυτή την περιοχή. Γιατί δεν είναι μόνο μια περιοχή που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι κεφαλαιώδης για όλη την ανθρωπότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής με την κλιματική αλλαγή θα ανοίξουν νέοι θαλάσσιοι δρόμοι, αλλά θα υπάρξουν και νέε απειλέ οι οποίε θα προκύψουν από την τήξη των πάγων τη Αρκτική. Υπάρχει λοιπόν μια όλο και πιο ταχεία τήξη των πάγων στην περιοχή της ακτική Πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν τεράστια η μάζα των πάγων της ακτική, αλλά εφέτος βλέπουμε με τι, τα τελευταία χρόνια μάλλον έχουμε δει με τι ταχύ ρυθμό έχει μειωθεί αυτή η κάλυψη πάγου της Αττικής. <clears throat> Μόνο το χειμώνα ξανακαλύπτεται όλη αυτή η περιοχή από τον πάγο, ενώ το καλοκαίρι όλο και περισσότερο δεν υπάρχουν πια δεν καλύπτεται πια από τον ε, πάγο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να σκεφτούμε καλύτερα και να επιβάλλουμε ένα γενικότερο μορατόριο για όλες τις δραστηριότητες μέσα στην ε, ακτική περιοχή που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το στρώμα πάγου εκεί. Δεν μιλώ για την ε, Βόρεια Σουηδία ή την Μόρια Φιλανδία εδώ πέρα, αλλά και για όλες τις άλλες περιοχές. Ξέρουμε ότι η εξόριξη πετρελαίου από υποθαλάσσια κοιτάσματα μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλα προβλήματα περιβάλλοντος. Έχουμε δει και στο παρελθόν φυσικές καταστροφές που προέκυψαν από ατυχήματα σε τέτοιες εξορίξεις πετρελαίου σε πιο θερμές θάλασσες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε αυτό το μορατόριο <clears throat> να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα ότι οικονομικά δεν είναι εκμεταλλεύσιμα αυτή τη στιγμή τα κοιτάσματα στην ε, Ακτική. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε καμία χρονική στιγμή δεν θα προχωρήσει κανείς σε εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων. Να υπάρξει λοιπόν ένα πραγματικό moratorium και είναι απαραίτητο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εστιάσει τις προσοχές, την προσοχή του στην προστασία της ε, περιοχής Αρκτικής. Θα πρέπει να καταλάβουμε και τις επιπτώσεις της αλλαγής το, της κατάστασης της ε, Αρκτικής για την κλιματική αλλαγή και για το επίπεδο των ωκεανών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος από τις έναντι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι που πήραν το λόγο πριν από μένα, η Αρκτική θέτει αυτή τη στιγμή δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι φυσικοί πόροι που βρίσκονται στην περιοχή αυτή μια περιοχή η οποία βρίσκεται λίγο εκτός των γεωπολιτικών μελημάτων και της διπλωματίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πετρελαίου που δεν έχει ακόμα τύχη εκμετάλλευση, ένα 30% περίπου φυσικού αερίου που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Όλα αυτά οδηγούν σε έναν πιθανό ανταγωνισμό εκμετάλλευση των πόρων αυτών και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και περισσότερε εντάσει. Και όπω είπαν και οι προλύσαντε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αφενό να τηρείται πλήρω το διεθνέ δίκαιο, αλλά και να διατηρήσουμε το status quo στην περιοχή. Μια περιοχή δηλαδή ειρηνική με χαμηλέ εντάσει και να αποφύγουμε πάση θυσία τη στρατιωτικοποίηση τη περιοχή αυτή. Παράλληλα όμως τίθεται και ένα άλλο πρόβλημα. Το ζήτημα της περιβαλλοντικής ζημίας που θα μπορούσε να πλήξει την περιοχή αυτή και το μοναδικό οικοσύστημα που έχει αυτή η περιοχή. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό κατ' επέκταση θα περάζει πάρα πολύ και τους τοπικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν είναι πολλοί, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και δεν θα πρέπει να τους ξεχνάμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό συντοποιώντας επίσης πόσο ο βόρειος αυτός διάδρομος γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες όπως και η Ιαπωνία που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προσπαθήσουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσουμε το θετικό πνεύμα συνεργασίας που υφίσταται ακόμα στην περιοχή και να προωθήσουμε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στις, ε, στην βιώσιμη ανάπτυξη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουμε την περιοχή αυτή σε περιβαλλοντική καταστροφή, σε μια αύξηση των κλιματικών φαινομένων που θα επηρέαζαν την όλη περιοχή πάρα πολύ αρνητικά. Στο ψήφισμα αυτό αναφερόμαστε σε κάποια σημεία στην χρηματοδότηση των υποδομών στην περιοχή. Θα θέλαμε εμείς να υποβάλουμε περισσότερες τροπολογίες στο σημείο αυτό λέγοντας ότι ναι μεν θέλουμε υποδομές αλλά θα πρέπει να έχουμε χρηματοδότηση υποδομών που θα επηρεάσουν αρνητικά την περιοχή αυτή. Δεν θα θέλαμε δηλαδή να έχουμε έρευνες επιστημονικές στην περιοχή αυτή, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια αρνητική οικονομική εκμετάλλευση των πόρων της περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σεβαστούμε αυτό προκειμένου να μην έχουμε ένταση ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μορατόριο τα επόμενα χρόνια, ελπίζοντας ότι στο πότερο μέλλον θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης το οποίο θα είναι βιώσιμο και ζητάμε και εμείς ε, όχι απλώς μείωση, αλλά παντελή εξάλληψη αρνητικών παραγόντων όπως ο μαύρος άνθρακας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντοπίσουμε ότι η πρόταση που γίνεται αυτή τη στιγμή για μια απλή μείωση δεν επαρκεί. Είναι πολύ σημαντικό να ζητήσουμε μια εξάλληψη του μαύρου αυτού άνθρακα, όπως άλλωστε έχει υποθεί πολλές φορές στο παρελθόν και από την ίδια την είπατε εκπρόσωπο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιακονσάρη έχει τώρα τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκιώδης Συγγετρία των Σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή Εξωτερικών και όπως οι συναδελφοί μου έτσι και εγώ θεωρώ ότι το σχέδιο αυτό είναι καλογραμμένο και ισορροπημένο είναι γεγονός αυτό το οποίο έχει ακουστεί αρκετές φορές ότι δηλαδή η συνεργασία στην Αρκτική είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε και την συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το Συμβούλιο της Αρκτικής έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και η συνεργασία συνολικά έχει αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο λοιπόν λείπει είναι οικοδόμηση συνεργασιών και όταν μιλάμε για την ε, βόρεια διάσταση Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία. Τα όσα έγιναν έχουν δημιουργήσει νέε εταιρικέ σχέσεις. Παραδείγματο χάρη η Ισλανδία, ο Καναδάς και άλλες χώρε είναι παρατηρητέ και καλωσορίζω το ότι ο ρόλο της Ρωσίας περιγράφεται με τρόπο ισορροπημένο στο κείμενο αυτό. Για τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ μίλησαν για το μορατόριο. Το ρωτήσαμε τους ντόπιου και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, νομίζω πως ε, το σκεφτικό αυτό του μορατόριου είναι πραγματικά δηλητήριο. Αυτοί το βλέπουν ως δηλητήριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνή κοινότητα πρέπει να δράσουν ε, με τρόπο παραδειγματικό. Πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε τους εθνικούς πόρους σεβόμενοι τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και ντόπιων λαών. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή στην οποία ζουν άνθρωποι. Δεν είναι ο νότιος πόλος, στην Αρκτική ζουν άνθρωποι. χρειάζονται ακριβώς τέτοιες υποδομές για να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους με τρόπο αηφόρο και να θυμόμαστε ότι η Αρκτική α, ανήκει και στην εσωτερική αγορά. Και χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για τηλεπικοινωνία, δρόμους, αεροδρόμια Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και όταν σκεφτόμαστε αυτές τις ε, προκλήσεις, ε, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την αηφόρο οικονομική ανάπτυξη. Είναι προβληματικά αυτά τα οποία αναφέρονται όμως στις παραγράφους 6 και 7. Οι προθέσεις είναι καλές, αλλά θέλουμε υποχρεωτική περιβαλλοντική αξιολόγηση των επενδύσεων. Ήδη τώρα τα κράτη της Αρκτικής κάνουν περιβαλλοντικές αξιολογήσεις. Και είναι κάπως προβληματικό να κάνουμε εμείς κήρυγμα σε Καναδούς ή Νορβηγούς ή Ισλανδούς ότι να τους πούμε ότι εσείς πρέπει να κάνετε καλύτερες αξιολογήσεις του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Ε, δηλαδή, ε, σαν να κάνουμε κήρυγμα. Ο μεγάλος αδερφός που λέει στους άλλους τι θα κάνουν. Πρέπει να έχουμε μάλλον κάποιες βέλτιστες πρακτικές ή κάποιον πίνακα, έτσι, βαθμολογίας, κάτι τέτοιο. και βεβαίως ε, και η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να παίξει ένα ρόλο εδώ και έτσι να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες ε, στην Αρκτική ε, θα γίνονται με τρόπο σωστό. Πριν από λίγο καιρό υπήρξε μια συνάντηση των βουλευτών της Αρκτικής που πρότειναν έναν δίκτυ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και νομίζω πως μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την ιδέα και σε αυτή την έκθεση. Οι συγητές μίλησαν για την εμπλοκή των ντόπιων στην ανάπτυξη της Αρκτικής. Και βεβαίως οι Σάμι είναι από τους αρχαιότερους αυτόχθονες ε, στην Ευρώπη. Θα έπρεπε να έχουν μια εκπροσώπηση στις ε, Βρυξέλλες. για να μπορούν ε, βεβαίως ε, να προωθούν τα συμφέροντά τους. Και εμείς ε, έχουμε προωθήσει αυτή την ιδέα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε μιλήσει για την σύσταση ενός κέντρου πληροφόρησης για την Αρκτική. Συνολικά λοιπόν είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική ιδέα. Ευχαριστώ και Σντόφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους συνεισηγητές μιλάμε για το περιβάλλον της Αρκτικής και πρέπει νομίζω να τονίσουμε την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ε, περαιτέρω προκλήσεις και στην αλλαγή του περιβάλλοντος. Και το συζητάμε με διάφορες χώρες ε, του Συμβουλίου της Αρκτικής, ε, Καναδά, Ρωσία, είπα και βεβαίως εν ώψη της συνεργασίας για την COP21, ε, ε, μετά την COP21 στο Παρίσι. Πρέπει και αυτό να το σεβαστούμε, αλλά βεβαίως να δούμε και τι γίνεται με τους κατοίκους σε μια Αρκτική, η οποία θα αναπτύσσεται. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα, ένας εθνικός δρυμός ή πάρκο. Πρέπει να μπορεί να αναπτυχθεί και να έχει και επιχειρήσεις και κάποιοι ζητάνε εργοστάσια. Και ξέρουμε πως θα υπάρξουν και νέοι ε, διαβλοί στην θάλασσα. Και το τι θα γίνει βεβαίως με την έρευνα και την διάσωση είναι επικίνδυνες οι περιοχές αυτές και Πρέπει επίσης να σκεφτούμε και πρέπει βεβαίως να συνεργαστούμε στενά με τους ε, γειτονές μας όπως η Ρωσία. Η Αρκτική είναι ένας τομέας και μια περιοχή όπου Έχουμε ήδη μία συνεργασία και πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στις περιοχές εκείνες που έχουν σημασία για την Αρκτική και όπου έχουμε κοινά συμφέροντα. Έχουμε λοιπόν φοβερά ε, οικονομικές δυνατότητες και για να προωθήσουμε βεβαίως την ειρηνική συνεργασία. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω. Ευχαριστώ. Κύριος Σλέκ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ την κυρία Πιτικάνη και τον κύριο Πατ, τους δύο εισηγητές για μια ιδιαίτερα καλά εξισορροπημένη έκθεση. Ε, χαίρομαι που σημειώνω ότι και από την πλευρά των εισηγητών και από την πλευρά της Κομισιόν υπογραμμίζεται ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής και της ε, αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Διότι οι αλλαγές του περιβάλλοντος που γίνονται στην περιοχή της Ακτικής προχωρούν με πιο ταχύ ρυθμό από ότι οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημασία που αποδίδεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέσα στη, στο σχέδιο Ιδίως την ιδέα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της Ακτικής θα πρέπει να σημαίνει και διατήρηση του τοπικού οικοσυστήματος και των τοπικών κοινωνιών. Από την άποψη αυτή, συμφωνώ απόλυτα και ενθαρρύνω την καλύτερη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες που έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτές τις κοινότητες για να αναπτύξουμε μια πλήρη και ενσωματωμένη στρατηγική. Το πιο σημαντικό επίσης είναι σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της περιοχής αυτής θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδος η οποία θα μπορέσει να γίνει σε διάφορες τομείς θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της βιωσιμότητας και το ε, εύθραυστο οικοσύστημα και οι θαγενείς πληθυσμοί να μην θυγούν από αυτήν την ανάπτυξη. Δεν πρέπει να υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο το ευάλωτο αυτό περιβάλλον της ακτικής. Χρειάζεται να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας οι καινοτομίε στην έρευνα είναι απαραίτητε για να διατηρηθεί η περιοχή τη Αρκτική, γι' αυτό πρέπει να ενθαρρύνουμε την επένδυση σε τέτοιε έρευνε. <clears throat> Επίση, πολύ σωστά, οι απορρίψει πετρελαίου, οι διαρροέ πετρελαίου με βαρέα κλάσματα έχουν θεωρηθεί ότι είναι σοβαρά προβλήματα για την περιοχή αυτή. Επομένω, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την ε, έρευνα και κοιτάσματα και τι μεταφορέ στην περιοχή. Σαφχάουζεν. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πανταχού παρούσα. Θέλει να τα κάνει όλα και για να μπορεί να τα πετύχει έτσι μόνη της αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει τι ρόλο παίζουν οι υπόλοιποι φορείς. Υπάρχει ήδη το Ακτικό Συμβούλιο με τη Δανία, την Σουηδία και την Νορβηγία, αλλά υπάρχουν και άλλα μέλη, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και τα λοιπά, που είναι παρατηρητέ στο Αρκτικό Συμβούλιο. Μα, συγγνώμη, τι προστιθέμενη αξία θα φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το να αναπτύξει μια τέτοια πολιτική τη στιγμή που ήδη οι ενδιαφερόμενε χώρε και οι μεγάλε ευρωπαϊκέ δυνάμει εμπλέκονται ήδη στο Αρκτικό Συμβούλιο. Επίσης, ποια είναι τα στρατηγικά ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αν το κείμενο είναι εξισορροπημένο, εδώ διαβλέπω ότι υπάρχει κάποια αιχμή κατά της Ρωσίας. Γιατί όταν μιλάμε για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φαίνεται πάντα να μας ενδιαφέρει ο ειρηνευτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολλές φορές και η αναμόχλευση αντιπαραθέσεων ως αισχυώδης λοιπόν εισηγητής από τη δική μου ομάδα. Θέλω να τα τονίσω όλα αυτά και πιστεύω ότι είναι περιττή η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο χώρο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος να λάβει το λόγο, μπορούμε να, ξαναδώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Φέλιξ Λίνιμαν, από την DG Environment. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ για την κοινή αυτή συνεδρίαση Άφετ και Ένβη. Εκτιμούμε πάρα πολύ το ότι από κοινού αποφασίσατε να συζητήσετε και να αξιολογήσετε την έκθεση αυτή και σας ευχαριστούμε και για το σχέδιο έκθεσης που έχει υποβληθεί από τους συνεισηγητές. Όπως γνωρίζετε, η κοινή ανακοίνωση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αστικά από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπάθησε πραγματικά να επικεντρωθεί στις διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που άπτονται της Αρκτικής. Εγώ θα ήθελα να αφαιρθώ στο διάλογο με τους γενείς πληθυσμού καθώς επίσης και να αναφερθώ στη δημιουργία ενός φόρουμ ενδιαφερομένων για την περιοχή της Αρκτικής. Στα πλαίσια του φόρουμ αυτού θα προσπαθήσουμε να ευθυγραμμίσουμε και να συντονίσουμε όλα τα μέσα και τις πολιτικές χρηματοδότης που χρησιμοποιούμε για την περιοχή της Αρκτικής ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε επίσης ότι προσπαθώντας να θεσπίσουμε και να δημιουργήσουμε το φόρουμ αυτό, ξεκίνησε μια διαβούλευση. Διαβούλευση η οποία θα πρέπει να μας βοηθήσει να κατευθύνουμε κάπως την ε, συνεισφορά που θα πρέπει να γίνει στο φόρουμ αυτό και προβλέπεται επίσης και μια σημαντική εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχει ο Επίτροπος Βέλλα, η Επίτροπος Βέλλα μάλλον, η ύπατη εκπρόσωπος, καθώς επίσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι και εκπρόσωποι της Φιλανδικής Προεδρίας του Αρκτικού Συμβουλίου. Αυτό θα γίνει το την ερχόμενη άνοιξη. Να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις για κάποιες από τις προτάσεις που διατυπώνονται στο σχέδιο έκθεσης. Αφενός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να λάβει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά αυτό το κέντρο το οποίο προτείνεται, κέντρο πληροφοριών όσον αφορά την περιοχή της Αρκτικής και θα θέλαμε επίσης να γνωρίσουμε πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί βιώσιμα ένα τέτοιο κέντρο πληροφοριών. Θα θέλαμε λοιπόν επ' αυτού περισσότερες πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφετέρου, εμείς συλλέγουμε αυτή τη στιγμή πληροφορίες για τη δημιουργία του φόρουμ αυτού για την αρκτική περιοχή και ήδη στις ιστοσελίδε μας υπάρχουν αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τις συνεξελίξει δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Αρκτικής Υπάρχουν δηλαδή ήδη διαθέσιμε πληροφορίε οι οποίε είναι προσβάσιμε. Και βέβαια διεξάγονται, όπω ξέρετε, και πολλέ μελέτε και πολλέ έρευνε για την περιοχή. Από την άλλη, θα μπορούσαμε όντω να θέσουμε κάποια ερωτήματα για την παράγραφο 6 και 7 του εγγράφου, όσον αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου, περιβαλλοντικού αντικτύπου, Όντω θα πρέπει να γίνει μια τέτοια νέα αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου και οποιαδήποτε τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ποια είναι επομένω η προστιθέμενη αξία τη ενισχυμένη διαδικασία περιβαλλοντικού αντικτύπου προτείνετε εσεί στην έκθεσή σα. Και καταλαβαίνετε ότι αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε ενδεχομένω η περιοχή τη Αρκτική να βρεθεί σε υποδέστερη θέση σε σχέση με άλλε περιοχέ για τι οποίε γίνονται τέτοιε μελέτε αντικτύπου. Δεν θα ήθελα τώρα να αναλώσω πάρα πολύ από το χρόνο σα και ενδεχομένω να πρέπει να δώσουμε το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Α ακούσουμε τώρα όντω τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, τον κύριο Τσέβιτ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι ε, καλωσορίζουμε οποιαδήποτε υποστήριξη θα μπορούσε να παράσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την διαδικασία αυτή δημιουργία μια ολοκληρωμένη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αρκτική. Ήδη από το 2008 έχουν γίνει σπουδαία πράγματα και θεωρώ ότι η επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων είναι πολύ σημαντική. Η κοινή ανακοίνωση σε καμία περίπτωση δεν είναι διεξοδική, δεν καλύπτει κάθε πιθανό ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να προκύψει στην περιοχή της Αρκτικής. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται στο κείμενο αυτό, αλλά αντικατοπτρίζονται στην παγκόσμια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι στα ζητήματα ασφάλεια. Η κοινή πάντω αυτή ανακοίνωση είναι ιδιαίτερα πλήρη για τα σημαντικότερα σημεία, τα κέρια σημεία, τα οποία θίξατε κι εσεί εδώ σήμερα. Προστασία του περιβάλλοντο, κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και διεθνή συνεργασία. Στους τομείς λοιπόν αυτούς, εμείς ε, έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συμβολή της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας. Και τονίσαμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ανθρώπων που κατοικούν την περιοχή αυτή και δι' των γηγενών πληθυσμών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι όντω το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευθυγραμμίζεται με τι προτεραιότητε που και εμεί εντοπίσαμε στην ακίνωσή μα. Όπω και ο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι και εγώ θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα όσον αφορά τι παραγράφου 6 και 7 του κειμένου. Η πρωτοβουλία που προτείνεται είναι σημαντική, σίγουρα. Αλλά ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συζητήσεις που γίνονται εδώ πέρα, αλλά και να κάνουμε κι εμείς περαιτέρω συζητήσεις για να δούμε αν τελικά όντως θα πρέπει να συσταθεί ή να δημιουργηθεί, μάλλον να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή την οποία προτείνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται για τις ε, διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες και αυτό συνάδει με τη δική μας την ανακοίνωση. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να επιμείνουμε στο ζήτημα της ε, έρευνας στον τομέα της Αρκτικής. Και με αυτό προφανώς συμφωνούμε και νομίζουμε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό θα μπορούσαμε να διαδραματίσουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πραγματικά συνιστά θέμενη αξία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για κοινοτικά προγράμματα έρευνας ε, στον τομέα αυτό. Προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ορίζοντα 2020 για παράδειγμα. Τέλος, από προσωπικής πλευράς θα ήθελα να γίνεται μία αναφορά στην βόρεια διάσταση, την οποία άλλωστε ανέφεραν και ορισμένοι ευρωβουλευτές στη σημερινή συζήτηση. Νομίζω ότι η βόρεια διάσταση είναι ένα πλαίσιο πολιτικής, στο οποίο συμμετέχει τόσο ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ρωσία, η Νορβηγία αλλά και η Ισλανδία. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνεται μία αναφορά και σε αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ας κλείσουμε τώρα τη συζήτηση δίνοντας πάλι το λόγο στον εισηγητή κύριο Πάιτ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλιά σας και αναμένω τις ε, τροπολογίες σας. Ε, μετά μαζί με την Σύρπα είναι τη συνεισηγήτρια και όλους τους σκιώδης συγητές θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε τελικά να υπάρξει μια ισορροπία και βεβαίως ταυτόχρονα και το βασικό σημείο αυτής της έκθεσης να παραμείνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδελφούς που έλαβαν μέρος στην συζήτηση και να θυμάστε πως οι προθεσμοί και τροπολογίες είναι 12 Δεκεμβρίου και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα είναι τροπολογίες στις 12 Ιανουαρίου και ψηφοφορία των δύο επιτροπών στις 31 Ιανουαρίου. Δίνω τον λόγο τώρα στον κύριο Μπρόκ για να κηρύξει την λήξη της ε, κοινή συνεδρίας. Σε ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Νομίζω πως έχουμε μια καλή βάση εδώ αν κατάλαβα καλά την συζήτηση. Δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που ε, μας ε, ενώνει, νομίζω, η προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, νομίζω. Το... Χαίρομαι για το ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Σας ευχαριστώ πολύ.